Έχουμε εδώ και εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών παρόντες που θα παρακολουθήσουν την ψηφοφορία. Καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ όλοι έτοιμοι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ωραία. Ας αρχίσουμε. Ψηφίζουμε τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε μετά από τις διοργανικές ε, συζητήσεις 11 του μηνός υπέρ παρακαλώ. Α, είναι ονομαστική, συγγνώμη. ένας παραπάνω από το EFF και ένας παραπάνω που τους σοσιαλιστές ψηφίζουν. Ωραία τώρα. Πέρας της φοφορίας. 38 ψήφοι υπέρ, 14 κατά και 2 αποχές. Ευχαριστώ κυρία Μωράν Σαρτιέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ψηφοφορία αυτή μοιάζει να μην είναι τίποτα. Στην πραγματικότητα όμως έχουμε πίσω μας 26 μήνες σκληρής δουλειάς. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την συνεισηγήτριά μου, την κυρία Άγνες Γιονγκέριους, η οποία δούλεψε πάρα πολύ και πολύ καλά μαζί με μένα και πολύ μας την ομάδα. Το Ρομπέρ επίσης από τη γραμματεία της Επιτροπής μας, θέλω να ευχαριστήσω. Φρασουά, Λάρα, Γιάν και Αλένα που είναι η πολιτική μας σύμβουλοι, λέω η πολιτική μας σύμβουλοι γιατί πραγματικά ήταν ε, μια ομαδική δουλειά αυτή που έγινε. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης το σύνολο της κοινοβουλευτική μας επιτροπής γιατί αυτή η ωραία πλειοψηφία στην οποία καταλήξαμε σήμερα δείχνει ότι αντικατοπτρίζουμε ακριβώς το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε, που είναι μιας κοινωνικής Ευρώπης, η οποία προστατεύει τους εργαζόμενους και η οποία στην εσωτερική αγορά μεταξύ των επιχειρήσεων φροντίζει να εγκαθιδρύσει έναν θεμητό ανταγωνισμό και ισορροπημένο. Εργαστήκαμε λοιπόν για να αποφύγουμε την κατάσταση που είχαμε στην αρχή και να αποφύγουμε το διχασμό ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Βλέπετε λοιπόν ότι με πολύ σκληρή δουλειά, ακούγοντας ένα τον άλλον, με διάλογο, τα καταφέραμε τελικά να βελτιώσουμε την οδηγία αυτή για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιονγκέριους. Δεν θα επαναλάβω όλα τα ονόματα αυτών που ευχαρίστησε η Ελίζαμπετ. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δράξω αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την ίδια την Ελίζαμπετ. Γιατί και εκείνη επένδυσε πάρα πολύ χρόνο, έβαλε ενέργεια, πνεύμα. Βοήθησε να γίνει καλά αυτή η δουλειά. Οπότε θα ήταν σωστό να σας ευχαριστήσουμε και εσάς, Ελίζαμπετ. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε ακόμα την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Αν τα καταφέρουμε, θα έχουμε αλλάξει κάτι προ όφελο των εργαζόμενων και προ όφελο των επιχειρήσεων εκείνων που θέλουν να παίξουν σωστά το παιχνίδι. Οπότε ευχαριστώ και εγώ όλους ε, όσους ευχαρίστησε η Ελιζαμπέτ και την ίδια επίσης προσωπικά. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και τις δυο σας. Δύο πολύ δυνατές γυναίκες. Συνεχίζουμε τώρα και θα ψηφίσουμε την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση υπέρ. Α, είναι ονομαστική βέβαια, ναι. Οπότε ψηφίστε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. 50 υπέρ, 4 κατά και καμία αποχή. Συνεχίζουμε. Πρόκειται για τις απαιτήσει εφαρμογής και τους ειδικούς κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών. Ο κατάλογος ψηφοφορίας συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 108. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τροπολογία 108. Τέλος της ψηφοφορίας. 21 ψηφί. υπέρ, 33 κατά. Απορρίφθηκε. Καμία αποχή. 106 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξω πάλι. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλος. 22 υπέρ, 31 κατά και μία αποχή. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 107 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε και την 107. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ. And the vote is now closed. Τέλος της ψηφοφορίας. 25 ψήφοι υπέρ, 30 κατά και καμία αποχή. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ τη συμβαστική 10. Τέλος της ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 32 κατά. Και μία αποχή. Απορρίφθηκε. Οπότε πάμε την εναλλακτική συμβιβαστική 10. Και πάλι ηλεκτρονικά όμως να ψηφίσουμε καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ. Εναλλακτική συμβαστική 10. Τέλος. 43 ψηφί υπέρ, 11 κατά και μία αποχή. 115 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την τροπολογία 115. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλος. 24 υπέρ, 26 κατά και 5 αποχές. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Καλώς. Ελέγχουμε για την 116 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. 28-27. Και κάμια αποχή. 122 τώρα. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. 122. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίστε. Τέλος. «28 κατά και 27 υπέρ και καμία αποχή». Τροπολογία 117 υπέρ, Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την 117. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. «23 υπέρ, 32 κατά». Απορρίπτεται. 119 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πιστεύω. 118. Να ελέγξουμε την 119 θέλετε. Ωραία, ηλεκτρονικά, 119. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 34 κατά. 118 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 118. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 38 κατά, 17 υπέρ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Πολλές από τις ψηφοφορίες έχουν ε, ένα αποτέλεσμα πολύ τσιματσίμα. μα. θα ψηφίσουμε όλα ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι θα πάει πολύ πιο γρήγορα η ψηφοφορία. Αν ε, συμφωνεί η πλειοψηφία, ναι, να το κάνουμε. Θα το εκτιμήσουμε. 121 τώρα. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίφθηκε. 32 κατά. 22 120 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Με 48 ψήφους κατά. Τροπολογία 123. Ψηφίστε. Πέρασε. Απορρίφθηκε με 30 ψήφους κατά. 125. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με 32 κατά. Τροπολογία 124. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορριφθήκε με 45 ψήφους κατά. Τροπολογία 126. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε με 30 ψήφους κατά. Τροπολογία 127. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 31 ψήφι υπέρ. Τροπολογία 128. Καταπίπτει. Τροπολογία 129. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 41 ψήφι υπέρ. Τροπολογία 131. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της φοφορίας Απορρίφθηκε 26 ψήφοι κατά. Τροπολογία 130. 132. Μπορείτε να ψηφίσετε την 132. Τέλος της φοφορίας Εγκρίθηκε. Τροπολογία 133. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 10, 134, 135, 136 και 137 που είναι ίδιες. Τις ψηφίζουμε μαζί λοιπόν. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 138 τώρα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Απορρίφθηκε 48 ψηφικατά. 139 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 140. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Απορριφθήκε με 47 κατά. Τροπολογία 141. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε με 47 κατά. 142 τώρα. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 143. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 144. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 145. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 146. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Παρακαλώ κύριε Μαρτά. Ναι, σε αντίθεση με αυτό που υπόθηκε πριν, νομίζω ότι όταν πρόκειται για τροπολογίες του ENF μπορείτε να ζητήσετε ψηφοφορία διανατάσσεως της χειρός. Θα πάει πιο γρήγορα. Γιατί εδώ υπάρχει μεγάλη δημοκρατία. Φαίνεται, έτσι δεν είναι. Ολοφάνερο. Ωραία. 147 τώρα. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίφθηκε. 148 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στην τροπολογία 149. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 150. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 151. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε με 30 υπέρ. 152 έχει αποσυρθεί. Οπότε πάμε στην τροπολογία 153. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 11. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 34 ψήφοι υπέρ. Συμβιβαστική 13. Ψηφίστε παρακαλώ τη συμβαστική 13. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με 33, 32 συγνώμη, ψήφους κατά. Οπότε ερχόμαστε στο εναλλακτικό συμβιβαστικό 12. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβιβαστική εναλλακτική τροπολογία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίθηκε με 33 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική εναλλακτική τροπολογία 13. Τώρα μπορείτε να ψηφίσετε την εναλλακτική συμβιβαστική πρόταση 13. Τέλος. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. Συνεπώς, πρέπει να Ψηφίσουμε τροπολογία 199 τώρα. 199. Okay. You find it on page 14. Σελίδα 14. Για να δω γιατί και εγώ πρέπει να το βρω. 199. Εντάξει, φτάσατε. Μπορείτε να ψηφίσετε την τροπολογία 199. Σελίδα 14 στον κατάλογο ψηφοφοριών. Ναι. Εντάξει, ψηφίσατε όλοι για την 199. Παρακαλώ. Για την τροπολογία 199 έχουμε τη συμβαστική 15. Θα την ψηφίσουμε ή όχι. Ψηφίζουμε την τροπολογία 199. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Γι' αυτό δεν υπάρχει και αυτό που λέτε. «199» στη σελίδα 14 σας είπα. Εκεί είμαστε επειδή οι προηγούμενες όλες τροπολογίες έχουν καταπέσει. Παρακαλώ κύριε Γιονγκέριους. Όχι. Εσείς, παρακαλώ. Είπα ότι η συμβαστική 15 δεν καταπίπτει. Πρόκειται για κάτι διαφορετικό από την συμβαστική 13 που εγκρίθηκε το εναλλακτικό, εναλλακτική συμβαστική πρόταση. Η ε, κυρία Κιονγκέριου, δεν συμφωνώ πάντα με την ε, συνάδελφο Ντανούτα, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση έχει δίκιο. Γιατί είχαμε την εναλλακτική συμβαστική πρόταση 13, αλλά όχι τη 15. Αυτή θα πρέπει να ψηφιστεί. Γιατί αλλιώ ε, κάνετε μάλλον λάθος. Για ξανασκεφτείτε το, Πρόεδρε. Okay. Ε, I owe ε, οφείλω κάτι στην κυρία Γεσεβίκα. Εργότερα. Ένα λουλούδι, κάτι τέλος πάντων θα τις προσφέρω. Ευχαριστώ κύριε Σβέκα. Πάντως έχετε δίκιο. Οπότε θα ψηφίσουμε τώρα τη συμβιβαστική 15 που είναι στη σελίδα 14. Μα υπάρχει μια παρεξήγηση ίσως επειδή είναι παρουσιασμένα τα πράγματα έτσι όπως είναι παρουσιασμένα, αλλά εγώ πιστεύω ότι 15 δεν πρέπει να ψηφιστεί, γιατί καλύπτονται οι τροπολογίες αυτές από την 12. Ωραία. Μια στιγμή. Ψυχραιμία. Θα το χειριστούμε. Λοιπόν, και πάλι αλλάξαμε γνώμη, η κυρία Γιωσοβέκα. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία 199. Γιατί έχει ήδη καλυφθεί η συμβαστική 15 όταν ψηφίσαμε πριν από λίγο. Με το καμποτάζ. Τροπολογία λοιπόν 199 τώρα. Πρέπει να ψηφίσουμε τη 15, εγώ είμαι εισηγήτρια. Πρέπει να ψηφίσουμε τη 15. Δεν μπορώ να σας πιστέψω γιατί οι, οι δικοί μας εδώ πέρα λένε πως όχι. Πως δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τη συμβαστική 15 αφού έχει καλυφθεί το καμποτάζ. Οπότε θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 199. Λοιπόν, ψηφίστε παρακαλώ για την 199 ηλεκτρονικά. Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην ψηφοφορία, ψηφίστε τώρα για την 199. Μπορείτε να ψηφίσετε, ναι. Τι, δεν δουλεύουν τα μηχανήματα. Α, τώρα δουλεύουν, εντάξει. Ψηφίστε. 199 τροπολογία. Ένας παραπάνω ψηφίζει από το ΕΛΚ. Να βγει μια κάρτα. Ωραία. 31 ψηφί υπέρ, 20 κατά είναι το αποτέλεσμα για την 199. Παρακαλώ κύριε Μπέκερ. Συγγνώμη που σας ενοχλώ και πάλι όλους, όμως το σχόλιο στις παρατηρήσεις στη συμβαστική 15 λέει καταπίπτει αν το εναλλακτικό 13 εγκριθεί. Δεν εγκρίθηκε όμως. Δεν εγκρίθηκε. Και καταπίπτει μόνο αν έχει εγκριθεί το 13. Κάτι που δεν έγινε. Αν δείτε την εναλλακτική συμβιβαστική 13, θα δείτε ότι δεν εγκρίθηκε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρόεδρος, το πρόβλημα είναι η ασφαλμένη πληροφορία. Το ένα ήταν το καμποτάστο, το άλλο ήταν κάτι άλλο. Καλώς. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάντως για ε, τις προσπάθειές σας να βοηθήσετε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λοιπόν, 8β τώρα, σεβαστική 8β, σωστά. Ωραία. Ξαναμπήκαμε στη γραμμή μας. Μπορείτε να ψηφίσετε. Συμβαστική 8β. Τέλος της φοφορίας. Απορρίφθηκε με 33 κατά. Οπότε ψηφίζουμε την αναλλακτική συμβιβαστική τροπολογία 16, λέει ο πρόεδρος. Α, όχι. Τροπολογία 236. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τροπολογία 236. Κυρία Πρόεδρε, εάν καταπίπτει μια συμβαστική, τότε πρέπει να ψηφίσουμε τις τροπολογίες που υποτίθεται ότι καλύπτει αυτή η συμβαστική. Άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 200 τώρα. Sorry, we have to vote. Συγγνώμη. Εφόσον το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της συμβαστικής 8β ήταν αρνητικό, Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 200 τώρα. Μπορείτε να ψηφίσετε τροπολογία 200. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 239. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. 14. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 240. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. και απορρίφθηκε με 41 ψήφους κατά. Τώρα τροπολογία 236. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 28 κατά 26 υπέρ. Κύριε Κιονγκέριου, ζητήσα το λόγο. Α, όχι. Τροπολογία 205 τώρα με την τροπολογία 243 μαζί. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 241. Ψηφίστε. Τέλος της προφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 242 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Εναλλακτική συμβιβαστική 16 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε με 31 ψήφους. Πάμε στη σελίδα 23 λοιπόν. Και στην τροπολογία 333. Σελίδα 23 τροπολογία 333. Μπορείτε να ψηφίσετε τώρα. Τέλος της ψηφοφορίας για την 333. Και εγκρίθηκε με 33 ψήφους. 334 τώρα. Καταπίπτει. Οπότε πάμε στην τροπολογία 332. Μπορείτε να ψηφίσετε για την 332 παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με 30 ψήφους. Τροπολογία 335 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 336. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 28 ψηφί υπέρ, 27 κατά. Η επόμενη καταπίτη. Και πάμε στην τροπολογία 338 μαζί με την τροπολογία 339. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της φοφορίας. Εγκρίθηκε με 32 ψήφους. 340 τώρα. Καταπίπτει. 342 επίσης καταπίπτει. 341 και 343 επίσης καταπίπτουν. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 344. Μπορείτε να ψηφίσετε τώρα. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με 35 ψήφους. Τροπολογία 345 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 37 ψηφί υπέρ. Τροπολογία 346. Ψηφίστε. Τέλος. Παρακαλώ, κυρία Γιαστροβέκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως να υπάρχει ένα λάθος στον κατάλογο ψηφοφορίας μου, αλλά Έχουμε 345, 346, 300 που απορρίπτονται, έτσι λέει, rejected λέει δίπλα. Οπότε γιατί τις ψηφίσαμε. Δεν καταλαβαίνω. Είχαν ήδη απορριφθεί. Οπότε γιατί τις ψηφίσαμε. They were not rejected. They fell. Okay. Uh, we proceed with the uh, voting on amendment. 347 τώρα. Ε, μπορείτε να ψηφίσετε. The vote is open on 347. Τέλος της ψηφοφορίας τώρα. Εγκρίθηκε με 35 ψήφους.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 Λοιπόν, η γραμματεία μας σας δικαίωσε τώρα, κύριε Γιασκεβέκα, που σημαίνει ότι 344, 345 και 346 όντως δεν ψηφίζονται αφού έχουν απορριφθεί. Γι' αυτό πάμε στην 347. Μπορείτε να ψηφίσετε. Α, την ψηφίσαμε και εγκρίθηκε. Ωραία. Άρα πάμε στην 348 τώρα. Που καταπίπτει. Ε, ή όχι. Καταπίπτει η 348. Η 349 λέει no vote, δεν την ψηφίζουμε, άρα ψηφίζουμε την 350 τώρα. Μαζί με την 353. Μπορείτε να ψηφίσετε τώρα. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με 47 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 351 τώρα. Μαζί με την 354. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με 37 υπέρ. Τροπολογία 355 τώρα. Την ψηφίσουμε ή όχι. Όχι. 352 του κύριου Σίστερ. Μπορείτε να ψηφίσετε τώρα. 352. Τέλος της φοφορίας. Εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ. Η 355 όμως <clears throat> καταπίπτει. Συνεχίζουμε. Τροπολογία 357. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Απορρίφθηκε με 49 ψήφους κατά. Άρθρο 4. Πρόταση της Επιτροπής. Συμβιβαστική 17. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της φοφορίας. Απορρίφθηκε με 30 ψήφους κατά. Οπότε πάμε στην αναλλακτική συμβαστική 17. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της φοφορίας. Εγκρίθηκε με 36 ψήφους υπέρ. Τώρα, τροπολογία 300. 60 και 361. Όχι, καταπίπτουν. 362. Μαζί με την 363, επειδή είναι οι ίδιες και την 364. Μαζί λοιπόν αυτές οι τρεις τροπολογίες. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτονται με 35 ψήφους κατά. Τροπολογία 21 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 365. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε με 32 ψήφους υπέρ. Τροπολογία α, καταπίπτει. Και 22 και 366. Οπότε ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 367. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Ισοψηφία, αλλά απορρίπτεται τότε. Τροπολογία 23 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε με μία ψηφοδιαφορά. Συμβιβαστική αριθμός 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 28 τώρα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε με 30 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 30. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με 38 ψήφους κατά. Τροπολογία 29. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε με 32 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική τώρα αριθμός 2. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε Τροπολογία 32. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική 3 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε με δύο ψήφους διαφορά. Συμβιβαστική 4 τώρα μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίνεται με 38 ψήφους. Σαράντα ένα τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε με 45 υπέρ. Τροπολογία 42. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με 39 κατά. Τροπολογία 43. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε με 46. Συμβιβαστική 4α τώρα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της φοφορίας. Απορρίφθηκε με 33 ψήφους κατά. Ε, εναλλακτική συμβαστική 4α τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. και εγκρίθηκε με 38 υπέρ. Τροπολογία 46 τώρα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε με 42 ψήφους υπέρ. 47 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 49. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Με 29 κατά. Τροπολογία 48 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε με 46 ψήφους κατά. Τροπολογία 50. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε με 31 ψήφους υπέρ. 52 τώρα. 52 καταπίπτει. Μη 51 καταπίπτει. Και πάμε στην τροπολογία 53 που μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της οφόριας. Εγκρίθηκε. Με 41 υπέρ. Τροπολογία 54 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. εγκρίθηκε με 35 ψήφους υπέρ. Η 55 καταπίπτει. Η 56 καταπίπτει. 57 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ για την 57. Τέλος της προφορίας. 46 ψήφοι υπέρ. Συμβαστική 4β υπέρ. Μάλλον ψηφίστε ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίθηκε. Με 34 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 65 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Α, όχι, διορθώνει η Πρόεδρος. Με μία ψήφο διαφορά απορρίφθηκε. Τροπολογία 5. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 72. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. 69 τώρα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Και εγκρίθηκε. 29-26. Τροπολογία 71 τώρα. Α, καταπίπτει. Και η τροπολογία 79 καταπίπτει και 74. Όλες οι επόμενες καταπίπτουν μέχρι τη συμβαστική 5 στη σελίδα 33. Μπορείτε να ψηφίσετε λοιπόν για τη συμβαστική 5 τώρα. Τέλος της ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε με 32 υπέρ. Συνεπώ καταπίπτουν το 85 και πάμε στη συμβαστική 7. Μπορείτε να ψηφίσετε για τη συμβαστική 7. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με 34 υπέρ. Αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 96. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ. 97 τώρα. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε με 46 κατά. 98. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε, μάλλον απορρίφθηκε διορθώνει πρόεδρος, 30 ψήφοι κατά. Και η τροπολογία 99. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας για την 99 εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ. Και τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία για την τροποποιημένη έτσι γνωμοδότηση με ονομαστική ψηφοφορία, οπότε μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Έληξη ψηφοφορία, ναι. Και εγκρίθηκε. 30 ψήφοι υπέρ. 22 κατά και 2 αποχές. Παρακαλώ, κυρία Σεβιέκα. Μια στιγμή, μια στιγμή, γιατί δεν σας ακούω. Ναι. Ευχαριστώ. Δεν ε, άλλαξε απόψή μου. Να ξέρετε ότι καταψήφισα εγώ. Δεν καταγράφηκε μάλλον στο μηχάνημα η ψήφος μου. Καταψήφισα να ξέρετε. Συνεπώς 23 κατά αντί για 22 με τη δικιά σας ψήφο. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζοβέκα για την ε, βοήθειά σας ώστε να ψηφίσουμε καλά και σας ευχαριστώ όλους. Ήταν μια πολύ περίπλοκη ψηφοφορία αυτή, είναι αλήθεια. Ήταν ε, και ο κατάλογος ψηφοφορίας περίπλοκος, οι συμβαστικές. Ε, πολλοί από εσά βοήθησαν με τις παρεμβάσεις τους που ήξεραν πώς να ψηφίσουμε. Πάντως σας ευχαριστώ όλους γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, η ψηφοφορία η σημερινή και το συγκεκριμένο θέμα έχει τεράστια σημασία. Ωραία. Οπότε τώρα έχουμε προφερμανθεί και μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη περίπλοκη ψηφοφορία. Σημείο 12. Βοηθήστε μας και εδώ παρακαλώ για να προχωρήσει ομαλά η ψηφοφορία. Ας ε, προχωρήσουμε λοιπόν ώστε να μπορέσουμε να το διεκπαιρεώσουμε σωστά. Ξεκινάμε με τη συμβιβαστική 10. Λοιπόν, διανατάσεις της ισχυρός αυτή τη φορά. Συμβιβαστική 10. Αγαπητοί ε, Πρόεδρε, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε για άλλη μια φορά για ποιο θέμα ε, ψηφίζουμε, ε, διότι στη σειρά που έχω εγώ ξεκινούσαμε κανονικά με τη συμβιβαστική 8. Ε, κύριε Πρόεδρε, έχουμε ξυπνήσει όλοι. Yes, we are voting on George Bach's ε, ψηφίζουμε στην έκθεση του Ζόσμπαχ. Ε, και ψηφίζουμε στην ε, συμβιβαστική 10 υπέρ κατά υπέρ λοιπόν εγκρίνεται και Πηγαίνουμε στην σελίδα 2, στη συμβιβαστική 11. Άρχεται η ψήφο. Όχι. Θα το προσπαθήσουμε με ένα της χειρός. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 13α υπέρ κατά πιστεύω πρέπει να ελέγξουμε τη συμβιβαστική 13α για να είμαστε σίγουροι άρχεται η υποψηφοφορία για την 13α συμβιβαστική όταν δεν σηκώνετε τα χέρια σας πρέπει να κάνουμε ψηφοφορία έλεγχο Ψηφίσατε τη 13α. Πέρας. Εγκρίνεται με 46 ψήφους. Ναι, αλλά πρέπει να σηκώνει το χέρι. Πάμε στην τροπολογία 88, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 89, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε στη συμβιβαστική 14 υπέρ κατά θα ελέγξουμε τη συμβιβαστική 14. Ας ξαναπροσπαθήσουμε με ένα χειρός 14. Υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και πάμε τώρα στη σελίδα 10 στην τροπολογία 122 Όχι. Την 1.23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε την 124 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται με 41 ψήφους. Πάμε στην 125 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Οπότε πάμε στη σελίδα 13. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 15. Πάμε στη σελίδα 16 και την ε, τροπολογία 155 υπέρ κατά ε, ελέγχουμε την 155 πέρας εγκρίθηκε με 29 ε, ψήφους συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 160 υπέρ κατά απορρίπτεται 161 υπέρ κατά θα την ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία 161 τροπολογία πέρας απορρίπτεται με 40 ψήφους, 162 ε, έχει αποσυρθεί, οπότε πάμε στην 163 υπέρ, κατά, ε, ας ελέγξουμε την 163, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, καταπίπτει με 32 ψήφους 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 ε, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά θα ελέγξουμε την τροπολογία 168 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με 40 ψήφους. Ε, πηγαίνουμε τώρα στη συμβαστική 18. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε τη συμβαστική 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίθηκε με 33 ψήφους. Πηγαίνουμε στη συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 181 υπέρ κατά απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά ελέγχουμε την τροπολογία 182 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίθηκε με 27 ψήφους. Ψηφίζουμε την 1.83 υπέρ, κατά, αποχές πιστεύω ότι απορρίφθηκε, αλλά σε ελέγξουμε την τροπολογία 183, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίθηκε με 26 ψήφους, μία παραπάνω, 184 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε την 184, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίθηκε με τρεις ψήφους. Παρακαλώ κύριο Σιλκιώτης. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 3 υπέρ Συγγνώμη, τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 4, τροπολογία 26. Ε, ψηφίζουμε την 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, ελέγχουμε την τροπολογία 27, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, και εγκρίνεται με 29 ψήφους, τροπολογία 27, υπέρ, κατά, εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 44 ψηφίζουμε την τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη 8α υπέρ τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά θα ελέγξουμε την τροπολογία 49 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίφθηκε με 34 ψήφους. Ε, συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 στη σελίδα 25. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 71, υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε την τροπολογία 71, άρχεται η ψηφορία. πέρας και απορρίφθηκε με 28 ψήφους. Τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τέλος ε, ψηφίζουμε επί το συνόλου ε, του κειμένου μετά τις τροπολογίες, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και έχει εγκριθεί με 32 ψήφους, 14 κατά και 7 αποχές.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 że jeden raport głosujemy imiennie, drugi raport głosujemy przez podniesienie ręki. Yes, it can be complicated when we when we move from one. My my, I want to be reach the right result, so I'm sure that every vote is counted. And yes, there are more complicated voting lists and those who are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 Μπορείτε να μην δίνετε τον αριθμό της σελίδα, γιατί δεν έχουμε όλη την ίδια κατάλογο ψηφοφορίας και άρα δεν αντιστοιχεί στις ίδιες σελίδες. Καλύτερα μόνο τον αριθμό της τροπολογίας. Ευχαριστώ. I'll try to not... Θα προσπαθήσω εφεξής να μην το κάνω. Πάμε στην συμβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίθηκε με 51 ψήφους. Οπότε συνεχίζουμε στην τροπολογία 156 άρχεται η ψηφορία πέρας για την 156 και απορρίφθηκε για δύο ψήφους συμβιβαστική 11 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίφθηκε για 6 ψήφους. Εναλλακτική συμβαστική 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίθηκε με 43 ψήφους. Πάμε στην εναλλακτική συμβιβαστική 13. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε με 33 ε, ψήφους. Και πάμε στην τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. 166. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίθηκε με 29 ψήφους 167 άρχιτη ψηφορία πέρας και εγκρίθηκε με 29 ψήφους τροπολογία 169 και 168 ταυτόσημες και τις ψηφίζουμε από κοινού. Άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε με 30 ψήφους. Πάμε τώρα στην Τροπολογία 172, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται με 44 ψήφους. Πάμε στην 173. Μόνο το δεύτερο τμήμα της 173. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Πάμε στην ενελεκτική συμβαστική 14. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίθηκε. Πάμε στην ε, τροπολογία 188. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέρας. Και απορρίπτεται. Τροπολογία 193. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται με 34 ψήφους η 194 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με 27 συνολικά ψήφους 195 άρχεται ψηφορία ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται η 196 άρχη του ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται η 198 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Και εγκρίνεται με 40 ψήφους. Ε, πάμε στην 198. Έναρξη. Πέρας. Και απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται 199 καταπίπτει οπότε πάμε στην 200 άρχεται ψηφοφορία πες καταπίπτει ή 201 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται με 31 ψήφους 202 άρχιτη ψηφοφορία πέρας και απορρίπτεται η 203 άρχεται πέρας και απορρίπτεται. Οι 204, 205 ταυτόσημες ψηφίζονται από κοινού. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 206. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 207. Καταπίπτει η 207, οπότε πάμε στην 102, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. και εγκρίνεται Τροπολογία 21, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Καταπίπτει 209, οπότε πάμε στην 2.10, ψηφίζουμε τη 2.10, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Η 2.11, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. και απορρίπτεται. Η 2.13 μαζί με την 2.14 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 2.15 καταπίπτει και η 2.12 οπότε πάμε στην τροπολογία 216 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 44 ψήφους. Κατά πίπτη 17 και 18, οπότε πάμε στην εναλλακτική συμβαστική 15α, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίθηκε με 33 ψήφους. είναι στην συμβιβαστική 15B, ε, Β, η ψηφοφορία. 15 Β. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 15 Β, άρχεται, πέρας. συνέχεια την 15 ε, Β. Έληξα με 31 ψήφους υπέρ, 16 κατά. Πάμε στην συμβιβαστική 14 λοιπόν. Καταπίπτει. Πάμε στην 2 35 τροπολογία. Τη βρήκατε. Τροπολογία 235 άρχη ψηφοφορία. Πέρας. και εγκρίθηκε με 35 ψήφους. Πάμε στην συμβαστική 15 γάμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίθηκε με 33 ψήφους. Και πάμε στην τροπολογία 245 Ψηφίζουμε τη 245, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Τροπολογία 246, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται με 53 ψήφους. Τροπολογία 248 Άρχεται ψηφορία. Πέρας για την 248. Τροπολογία 248 των Σάιμον Κρίστινσεν και άλλων. Καταπίπτει, καταπίπτει. Συμβιβαστική 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 50 ψήφοι υπέρ για την συμβαστική 16. Πάμε στην τροπολογία 254, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται με 29 ψήφους. τροπολογία 265 άρχεται η ψηφορία πέρας απορρίφθηκε Πάμε στην 266, άρχη της ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 267 άρχεται πέρας Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17. Άρχη ψηφοφόρια. Πέρας. Εγκρίνεται με 53 ψήφους. Τροπολογία 2.71. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Ε, ύστερα από αίτημα των σοσιαλιστών. Για το πρώτο τμήμα λήξη της ψηφοφορίας και εγκρίνεται με 38 ψήφους. Το δεύτερο τμήμα πέρας και απορρίπτεται με 31 ψήφους. Τροπολογία 272, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 28 ψήφους. Και πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 25, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται Εναλλακτική συμβαστική 1. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 2 της ε, κυρίας Φοντανιέ. Άρχεται ψηφορία. Πέρας πίπτη 35. Ε, πέρας της ψηφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Δεν ε, λειτουργήσε, οπότε θα ξαναδοκιμάσουμε. Τώρα λειτουργεί. Τροπολογία 36 και το αποτέλεσμα είναι πέρας και εγκρίνεται συμβιβαστική 2 του ψηφορία πέρας εγκρίνεται εναλλακτική συμβιβαστική 3 του ψηφορία πέρας εγκρίνεται συμβιβαστική 4 άρχεται η ψηφορία. και εγκρίνεται με 51 ψήφους Τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 56 Άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται με 47 ψήφου, συμβιβαστική 5, άρχεται ψηφορία, πέρας, εγκρίνεται με 50 ψήφου. τροπολογία 63, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται 64 του ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται συμβιβαστική 6 πέρας της ψηφορίας εγκρίνεται με 50 ψήφους Τροπολογία 71. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται η 72. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται με 43 ψήφους. Τροπολογία 73 καταπίπτει, οπότε πάμε στην συμβιβαστική 7. Ο κύριος Μοντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα οι υπηρεσίε να μου εξηγήσουν την συμβατή σημείωση με την τροπολογία 71. Εάν είναι δηλαδή συμβατή με την 71 πρέπει να το ψηφίσουμε μαζί. Δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε οπωσδήποτε εκ νέου να κάνουμε μια εξαιρετικά αρνητική ψήφο για μια τέτοια τροπολογία. Ε, η 73 συμπίπτει ε, με την 71 και καταπίπτει σε περίπτωση που εγκριθεί η 72 και αυτό το λόγο εκτός μικροφώνου είναι σύμφωνα με τον κανονισμό. Οπότε πηγαίνουμε στη συμβιβαστική 7, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 48 ψήφους. Και πηγαίνουμε στην εναλλακτική συμβιβαστική 7 α, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 31 ψήφους, εναλλακτική συμβιβαστική 7β, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 32 ψήφους. Τροπολογία 11. Ψηφίζουμε την 11, άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε με 34 ψήφους. Τροπολογία 95. Άρχεται ψηφορία. Πέρας και εγκρίνεται με 33 ψήφους. Τροπολογία 97, άρχιε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 49 ψήφους. Τροπολογία 98, άρχιε ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται με 51 ψήφους. Ε, ε, η 98 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 41 ψήφους. Τροπολογία 100. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται για μία ψήφο. 101 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζει ένας παραπάνω από το EPP. Πάλι ένας πλεονάζων. και απορρίπτεται με 37 ψήφους. Ψηφίζουμε την τροπολογία 12, άρχεται ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε επί, το, επί του συνόλου του κειμένου, όπως έχει τροπολογηθεί. Πέρας της ψηφορίας. Έχετε ψηφίσει όλοι. Ωραία. Πέρας. Και εγκρίνεται με 31 ψήφους. It's Φίλοι μου, να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ε, ψηφοφορία. Αλλά τώρα θα ήθελα, όσοι δεν θέλετε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση στο επόμενο σημείο της Μύρισης διάταξης, να εξέλθετε τις αιθούσεις. Μπορείτε φυσικά ωραιότατα να παραμείνετε αν θέλετε να ακούσετε τον προσκεκλημένο μας, αλλά όχι να συζητάτε μεταξύ σας. Συνεχίζουμε με την ε, τακτική μας συνεδρίαση μετά από την ε, πάση των ψηφοφοριών. Επόμενο σημείο είναι η αξιολόγηση των οργανισμών υπό την εντολή ε, της ε, Επιτροπής, την μάλλον, της Επιτροπής Απασχόλησης. Θα δώσω το λόγο στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Γιώστ Κόρτε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να μας ενημερώσετε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαρά μου να βρίσκομαι εδώ απόψε για να σας προβάλλω τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης των ευρωπαϊκών οργανισμών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της δικής μου γενικής διεύθυνσης. Μιλάμε για το Eurofound στο Λονδίνο, σε DeFop στη Θεσσαλονίκη, το ETF στο Τωρίνο και την όσα στο Μπιλμπάου. Οι οργανισμοί αυτοί είναι διαφορετικοί, μεταξύ τους, αλλά είναι σημαντικό να εξετάζουμε πού και πού την απόδοσή τους. Γι' αυτό και ζητήσαμε μια εξωτερική ε, αξιολόγηση για να δούμε τις, ε, τις επιδόσεις τους. Σας παρουσιάσω σύντομα τα αποτελέσματα, γιατί θα πρέπει ίσως να δώσουμε και μια ευρύτερη εικόνα του πλαισίου στο οποίο συμβαίνουν όλα αυτά. Υπάρχουν ε, τρεις σημαντικές διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει και θα πρέπει να συγχαίονται γιατί είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να ακούσετε από την πλευρά μου ότι αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται. Πρώτη διαδικασία λοιπόν που έχει ξεκινήσει, που έχει γίνει μάλλον, είναι αυτή η ανάλυση αξιολόγησης που κάναμε. Ξεκίνησε αυτόνομα το 2015 και οι αξιολογητές ολοκλήρωσαν την εργασία τους νωρίτερα φέτος. Δεύτερον, χωριστά έχει ξεκινήσει μια διαδικασία τριμερούς διαλόγου για την αναθεώρηση των ιδιωτικών κανονισμών τριών εξ αυτών των οργανισμών. Πρώτο τριμερή διάλογο ήταν χτε μάλιστα και στόχο είναι να ευθυγραμμιστούν οι δυτικοί κανονισμοί στην κοινή προσέγγιση που συμφωνήθηκε ανάμεσα στους θεσμούς το 2012. Το πιο σημαντικό ίσως που συνέβη πρόσφατα είναι η πρόταση της Κομισιόν για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Περιεπασχόλησης. Δημιουργήσε δηλαδή μια ένα πέμπτο οργανισμό που πάλι εμπίπτει στις αρμοδιότητες της δικής σα Επιτροπής και, θα, και γι' αυτό θα κάνει η Μαρία Ματάης μια παρουσίαση που θα έρθει στην Επιτροπή σας στις 25 ε, Μαΐου. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν συνδέονται μεταξύ τους, αλλά δεν είναι, ε, ε, αλλά δεν είναι τα ίδια. Αξιολόγηση λοιπόν των ε, τεσσάρων οργανισμών. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο τα αποτελέσματα του εξωτερικού αξιολογητή. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή η γνώμη της Κομισιόν, είναι τα στοιχεία που πήραμε από τον εξωτερικό αξιολογητή BPMI ΕΚΟΗΣ που έχει σύμβαση για να κάνει αυτή, αυτό το έργο. Τι θα γίνει αφού λοιπόν θα σας έχουμε ακούσει και θα έχετε την ε, δυνατότητα κι εσείς να συμβάλλετε σε αυτήν ε, την υπό, τη διαδικασία. Θα συντάξουμε ένα έγγραφο εργασίας, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί ε, μετά τις θερινές διακοπές και από αυτού το έγγραφο εργασίας όπου θα περιλαμβάνεται και η δική μας αντίδραση σε αυτήν την εξωτερική αξιολόγηση, θα εργαστούμε. Επίση, θα κάνουμε ίσω και προτάσει για το ποιε ενέργειε ε, χρειάζονται ώστε να βελτιωθούν οι ε, επιδόσεις των οργανισμών. Αυτό θα το έχουμε, ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και σήμερα και αργότερα μέχρι ότου να ολοκληρωθεί η εκπόνηση αυτού του εγγράφου για να λάβουμε υπόψη για τι δικέ σα απόψει Το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή κλήθηκε να συμμετέχει σε ε, συνεντεύξει στη διάρκεια της αξιολόγησης. Φαντάζομαι πως ήρθαν σε επαφή με όλους σας και θα έχετε λάβει μάλιστα την έκθεση ολοκληρωμένη πριν από μια εβδομάδα. Σύντομα λοιπόν θα σας παρουσιάσω τα κύρια συμπεράσματα της εξωτερικής αυτής αξιολόγησης και αυτό που είναι σημαντικό είναι να εξετάσουμε τους τρεις άξονες που ζητήσαμε να αξιολογήσει ο ο ανεξάρτητος οργανισμός. Πρώτον, να δει ανεξάρτητα την ε, <coughs> αποτελεσματικότητα της επιδόσης και την προστιθέμενη αξία, καθώς και το ποια είναι η σκοπιμότητα ύπαρξη αυτών των οργανισμών. Ζητήσαμε να εξεταστούν οι συνδέσεις ανάμεσα σε αυτούς τους οργανισμούς, να εντοπιστούν οι δυνατότητες συνεργασίας. Ε, και στα εντολές τους. Επίσης τους ζητήσαμε να δουν στο μέλλον, δηλαδή ποια θα ήταν πιθανά σενάρια για το μέλλον αυτών των οργανισμών συμπεριλαμβανομένης της άφηξης της Ευρωπαϊκής Αρχής Απασχόλησης. Αυτοί ήταν οι τρεις άξονες όπου ζητήσαμε συγκεκριμένα να μελετήσουν ο αξιολογητής και είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε πριν σας παρουσιάσω σύντομα τα αποτελέσματα το πώς έγινε ακριβώς αυτό. Ο αξιολογητής εξέτασε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία έναντι των κανονικών και τυπικών έργων, εργασιών, καθηκόντων των οργανισμών. Δηλαδή, είδαν το καταστατικό, τι πρέπει να κάνουν αυτές οι, αυτοί οι οργανισμοί, είδαν τα προγράμματα εργασίας αυτών των οργανισμών και με βάση αυτό, ε, αυτά τα ε, ε, αναφορές αξιολόγησαν τους οργανισμούς. Δηλαδή δεν είναι πολιτική, πολιτικό εγχείρημα, ε, δηλαδή μήπως θα έπρεπε να δημιουργηθούν διαφορετικοί οργανισμοί, κάτι άλλο πολύ διαφορετικό. Οι δύο παλαιότεροι ε, χρονολογούνται από το 1975. 1975 έχουν τριμερή δομή, αλλά δεν ήταν αυτό το ερώτημα που θέσαμε. Πρόκειται για τεχνικής φύσης περισσότερο αξιολόγηση. Θέλω αυτό να το υπογραμμίσω, διότι δεν σκοπεύουμε εμεί ε, στην Κομισιόν με βάση αυτό το χαρτί, ε, αυτή τη μελέτη, να προχωρήσουμε σε σημαντική πολιτική πρωτοβουλία. Έχουμε λοιπόν μεμονωμένη εξολόγηση της ε, εφαπτώμενες δυνατότητες συνεργασίας και μετά το μέλλον. Για το πρώτο σημείο το συμπέρασμα είναι πολύ θετικό όσον αφορά την αποδοτικότητα ε, δηλαδή και τις επιδόσεις. Έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά, έχουν ε, ε, φέρει αποτελέσματα, έχουν επιτύχει τους στόχους που είχαν θέσει στα προγράμματα εργασίας και συνέβαλαν προς τους γενικούς τους στόχους. Εντοπίστηκαν κάποιες βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν για τις δημοσιονομικούς περιορισμούς, για καθυστερήσεις ε, στη ε, στα αποτελέσματα και κάποιες φορές η προσβασιμότητα και η αναγνωσιμότητα ε, των πορισμάτων δεν ήταν καλή. Και αυτό επανέρχεται στο θέμα της επικοινωνίας. Δηλαδή, πολλοί οργανισμοί από αυτούς δεν είναι ορατοί για τον κόσμο για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και για τους φορείς που λειτουργούν εδώ εντάξει, αλλά εκτός Ένωσης δεν είναι ορατά ε, τα επιτεύγματα και ε, τα αποτελέσματα, τα πορίσματα αυτών των οργανισμών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τέλος, χρειάζεται να εξετάσουμε πολύ εντατικά την ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων που θεσπίζουν οι ε, οργανισμοί με βάση τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Αυτές είναι που κατευθύνουν και τα προγράμματα εργασίας των οργανισμών. Και εκεί υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Παρόμοιο ε, συμπέρασμα όταν μιλάμε για αποτελεσματικότητα ε, υπάρχει μεγάλος, ε, μεγάλος βαθμός αποτελεσματικότητας παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και τους περιορισμούς σε ανθρώπινο δυναμικό. Η δομή για τα διοικητικά συμβούλια τριών των οργανισμών και εδώ μιλάμε για το Δουβλίνο, Eurofund, για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και την ΩΣΑ όπου έχουν διοικητικό συμβούλιο που είναι τριμερές, σημαίνει έχουν 87 μέλη έκαστος στο διοικητικό συμβούλιο και ο αξιολογητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό, αυτή η δομή έχει πολλά πλεονεκτήματα, αν και δεν συμμορφούνται απόλυτα και αυστηρά με την κοινή προσέγγιση. Αυτό αναφέρεται στην προσπάθεια που έγινε το 2012 για ευθυγράμμιση των οργανισμών. Το να διατηρηθεί η τριμερής ε, ε, δομή, ε, να διατηρηθεί η τριμερής αυτή δομή λοιπόν και γι' αυτό δεν τροποποιήσαμε. Δεν προτείνουμε τροποποίηση των ε, διοικητικών συμβουλίων των οργανισμών αυτών. Δεν θα το αλλάξουμε αυτό. Όταν ε, κανείς εξετάσει τις επιδόσεις, τα αποτελέσματα της υπηρεσίας που προσφέρουν και πάλι το συμπέρασμα είναι θετικό, και από την άποψη των ευρωπαϊκών θεσμών και από την άποψη των ενδιαφερομένων φορέων. Ωστόσο, οι περιορισμένοι πόροι δημιουργούν ε, και χάσμα ανάμεσα στο τι αναμένεται, στι προσδοκίε, στο τι περιμένουν τα κράτη-μέλη, κοινωνικοί και τα κράτη-μέλη και το τι μπορούν να προσφέρουν. Υπάρχουν βεβαίω περιορισμοί, αλλά δεν μπορούμε πάντοτε να απαντούμε στην. Ε, ε, στα αιτήματα λόγω των περιορισμών. Οι μοναδικοί συνδυασμοί ε, που προσφέρουν ε, αυτή η που προσφέρει ο τριμερής ε, χαρακτήρας των δομών αυτών είναι πολυθετική και αυτό είναι ένα πολυθετικό βέβαια συμπέρασμα. Τώρα, αυτό που είπαμε για τις εφαπτώμενες προοπτικές ε, και δυνατότητες συνεργασίας. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την αξιολόγηση της συνοχής της εργασίας των τεσσάρων αυτών οργανισμών και η αξιολόγηση εντοπίζει ότι υπάρχουν ε, ε, επικαλύψεις αν δούμε δηλαδή το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης, και οι δύο είναι αρμόδιοι για ε, την πολιτική κατάρτιση. Υπάρχει επικάλυψη. Στην πράξη δεν δημιουργεί δυσκολία γιατί έχουν διαφορετική επικράτη και φάσμα. Το Τωρίνο ασχολείται μόνο με τρίτε χώρε, ενώ το Σεντεφόπ τη Θεσσαλονίκη ασχολείται με τα κράτη-μέλη τη Ένωση. Ωστόσο, υπάρχει χώρο βελτίωση τη συνεργασία ανάμεσα στου οργανισμού, που σημαίνει ε, αυτή τη στιγμή είναι διμερής. Ε, ε, και αποτελείται από, μάλλον συνίσταται, σε ανταλλαγή γνώσεων και στοιχείων. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει μια πιο ουσιαστική συνεργασία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις μελλοντικέ προκλήσεις και εδώ ε, θα πρέπει και εμείς να παίξουμε κάποιο ρόλο στην Κομισιόν ώστε να ενθαρρύνουμε τους οργανισμούς αυτούς να βελτιώσουν το συντονισμό μεταξύ τους. Τέλος, ε, προοπτικές για το μέλλον. Μία ενδιαφέρουσα ερώτηση που έθεσαν οι αξιολογητές ήταν διάφορα σενάρια συγχωνεύσεως. Θα ήταν λογικό να συγχωνευθούν ίσως κάποιοι οργανισμοί, για παράδειγμα το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και το ETF ή το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και το Eurofund και ο αξιολογητής συμπεράνε τελικά πως ε, το γενικό κόστος και κίνδυνοι ε, μια συγχώνευσης ε, ξεπερνούν το, τα ωφέλη από μια συγχώνευση. Δηλαδή θα, δεν θα ήταν καλή ιδέα. Ακόμα και αν ο αξιολογητή όμω είχε φτάσει σε διαφορετικό συμπέρασμα, είναι σαφέ και το έχω αυτό συζητήσει με την Μαρία Τάισεν ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, τουλάχιστον σε αυτή τη θητεία, να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδου πρωτοβουλίε. Οπότε η Κομισιόν δεν θα ασχοληθεί με τέτοιο θέμα. Τώρα, υπό το φως των προκλήσεων και των κινδύνων που ε, περιλαμβάνονται στα διάφορα σενάρια συγχώνευσης, οι αξιολογητές συστήνουν ε, περισσότερο ένα πλαίσιο για ενισχυμένη συνεργασία. Εντάξει, είναι λίγο τώρα ευρωπαϊκή ορολογία, αλλά εσείς φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή σημαίνει ότι θα στηριχθεί καλύτερα η συνεργασία μεταξύ οργανισμών, και ε, θα είναι περισσότερο πολυμερής και ε, συνεργατική προσέγγιση. Τελευταία μου σχόλια για τις σχέσεις μεταξύ των υπαρχών των τετσάρων και του πέμπτου οργανισμού που θα στηθεί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Απασχόλησης, πράγμα το οποίο πρότεινε η Κομισιόν πριν από ένα μήνα. Εδώ οι αξιολογητές εξέτασαν κάπως πώς ε, αυτοί οι τέσσερις μπορούν να δουλέψουν μαζί. Η δυνατότητα, η πιθανή δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα στους τέσσερις και το νέο πέμπτο οργανισμό είναι περιορισμένη και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θα επανέλθει η Κομισιόν φαντάζομαι το Μάιο όταν θα παρουσιάσει την πρόταση και θα συζητήσει μαζί σας γιατί είναι πολύ διαφορετική οργανισμοί. Οι τέσσερις που ήδη υπάρχουν ε, κατά κύριο λόγο είναι προσανατολισμένοι στην έρευνα ενώ ο ΕΛΑ θα είναι, είναι επιχειρησιακό εργαλείο που θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν καλύτερα μεταξύ τους από ό,τι μέχρι σήμερα. Είναι δηλαδή μία δομή στήριξης. Δηλαδή ο νέος οργανισμός δεν έχει να κάνει με τις οργανισμούς που υπάρχουν ήδη περισσότερο. Με τη Eurojust ή με τη Europol θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε. Οι τομείς βέβαια είναι πολύ διαφορετική αλλά όσον αφορά τους στόχους, δηλαδή τη συγκέντρωση των εθνικών αρμοδίων σε μια ελαφριά δομή όπου μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα, και επίση ε, η παροχή καλύτερης ενημέρωσης στου ευρωπαίου πολίτε που θέλουν να εργαστούν και να διαμένουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Με την αξιολόγηση λοιπόν καταλήξαμε ότι δεν θα υπάρξει μεγάλος βαθμός συνεργασίας εκεί, αλλά Υπάρχει και μια ρήτρα ραντεβού που προβλέπει την αξιολόγηση της εντολής ε, των στόχων και των ε, αρμοθετήτων και καθηκόντων μετά από πέντε χρόνια. Θα έχουμε δηλαδή αυτόματα μια δυνατότητα πέντε χρόνια μετά από την έναρξη λειτουργίας του νέου οργανισμού να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε πώς θα έχει ε, λειτουργήσει και πάλι θα μπορέσουμε να ξανασυζητήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας με τους υπόλοιπους. Επί τη βάση αυτή τη αξιολόγηση λοιπόν και των πορισμάτων τη, αναλύουμε τι είδου συστάσει θα μπορούσαμε να ε, κάνουμε προ την Επιτροπή. Η συνέχεια που θα δοθεί θα λάβει υπόψη του δημοσιονομικού περιορισμού, καθώ και την ανάγκη να έχουμε περισσότερου περιορισμού κόστου. Το έγγραφο εργασία θα σα δοθεί μετά το καλοκαίρι και περιμένουμε την πολύτιμή σας συμβουλή και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε σε μια περίοδο που ασχολούμαστε περισσότερο από ποτέ με τους διάφορους οργανισμούς. Αρχίσαμε τριμερή διάλογο, έχουμε προετοιμαστεί, οπότε είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σαμπόν που ζήτησε το λόγο, την κυρία Σαντέρ μετά, κυρία Γιουγκέριος. Εντάξει, ωραία. Ο κύριος Σαμπόν, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέρφους που δέχονται να αλλάξει κάπως η σειρά γιατί πρέπει να μιλήσω για την αφαιρεγγιότητα με αυτούς που έρχονται από το Περσί, από το Παρίσι και δεν θα έπρεπε να τους αφήσω να περιμένουν. Ε, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ το Γενικό ε, Διευθυντή για τόσα είπε. Τώρα, εμείς όλοι μαζί δεν ήμασταν και τόσο εξαιρετικοί όσον αφορά αυτά που θέλουμε να κάνουμε και αυτά που θέλουμε να αποφύγουμε. Εμείς κάνουμε τον τριμερή μας διάλογο συγχρόνως με μία μελέτη η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και μετά συνεχίζουμε. Τέλος πάντων, προσπαθώ να καταλάβω ότι αυτά τα οποία τώρα μας είπατε, αναλύεται κτλ. είναι για το μέλλον. Έχουμε συζητήσει με τους συναδέρφους πριν ψηφίσουμε το κείμενο που τώρα συζητάμε στον τριμερή διάλογο. Εγώ ήμουνα, είμαι για το Eurofound εισηγητής και είναι ο οργανισμός αυτός που γνωρίζω εγώ καλύτερα. Πάντως, τι θέλω να πω. Στο δικό μας έργο προσπαθούμε να αποφύγουμε κάποια πράγματα. Η ιδέα μας είναι ότι οι οργανισμοί αυτοί, ή τέλο πάντων οι τρεις που γνωρίζω εγώ καλύτερα, Υπάρχει το Σέντεφοπ που κάνει πολύ καλή δουλειά. Από πριν, από τότε που ήταν στο Βερολίνο, έτσι. Μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ είμαι παλιό και τα ξέρω αυτά. Ε, με το Τωρίνο δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιες ε, διαιρέσει εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι οι δυνατότητε αυτών των οργανισμών ε, δεν, ε, είναι τέτοιες που δεν τι εκμεταλλευόμαστε όσο θα μπορούσαμε. Το είπατε κι εσείς και συμφωνώ μαζί σας. Ήμουν και 20 χρόνια στην ΟΚΕ. Δεν χρησιμοποιούμε αρκετά αυτούς τους οργανισμούς. Οι πελάτες τους δηλαδή, που θα έπρεπε η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, ε, και μπορεί να τους χρησιμοποιεί περισσότερο, τέλος πάντων, δεν τους χρησιμοποιούμε αρκετά αυτούς τους οργανισμούς που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και είναι κρίμα. Και στα άλλα θεσμικά όργανα, ίσως και στο Συμβούλιο, πάμε και εξοδεύουμε χρήματα και λέμε να κάνουμε μια εξαιρετική μελέτη σε δεν ξέρω εγώ τι, το κόστος των μεταναστών ή το gender gap ή ξέρω εγώ τι, ενώ τέτοιες μελέτες μπορούν να γίνουν καλύτερα στους οργανισμούς αυτούς και ακόμα χειρότερο μπορεί να έχουν ήδη γίνει από αυτούς τους οργανισμούς. Οπότε θα ήθελα να τους χρησιμοποιούμε περισσότερο, γιατί αν δεν τους χρησιμοποιούμε και αν καταλήξουν να έχουν ακαδημαϊκό μόνο κύρος, ε, θα τους μειώσουμε τον προπολογισμό κλπ. κλπ. Αυτή είναι μια πρώτη ιδέα μου για το μέλλον, έτσι, εντάξει. Δεύτερον, λίγο πολύ απαντήσατε βέβαια, θέλω να ακούσω και τους συναδέλφους. Πάντως εγώ δεν κατάλαβα ποτέ από πλευρά του Eurofound τουλάχιστον. Η νέα εργασιακή αρχή τι σχέσεις μπορεί να έχει με αυτά. Γιατί έχουμε ερευνητικά κέντρα, συμβουλευτικά κέντρα, αξιολόγησης. Τι σχέση έχουν αυτά με μία υπηρεσία που θα δημιουργήσει το, την εμβριακή κατάσταση ε, κανόνων εργασιακών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωραία, θα είναι οι επιθεωρητές, θα μας βοηθήσουν κτλ. Εντάξει, αλλά τα ερευνητικά κέντρα είναι κάτι άλλο. Και έχουν πολιτική διεύθυνση, δεν είναι πανεπιστήμια, εννοείται. Λέμε, έχουμε το πρόβλημα των μεταναστών. Λοιπόν, πείτε μας, τι γίνεται κάντε μια μελέτη για να μας δώσετε αυτή την απάντηση ή για τις ε, διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ή για οτιδήποτε άλλο. Ποια είναι η πραγματικότητα για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Δηλαδή, αυτοί οι οργανισμοί είναι οργανισμοί τους οποίους μπορούμε να συμβουλευτούμε για να μάθουμε την πραγματικότητα και να μην μένουμε στα λόγια και στις διαδόσεις. Αυτά. Ξέρω ότι και εσείς ε, συμφωνείτε αλλά αυτό ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όσον αφορά το μέλλον. Και θα ολοκληρώσω με κάτι που έχουμε ήδη συζητήσει. Έχει ήδη περάσει. Στηρίζω το κείμενο βεβαίως του Κοινοβουλίου. Εκεί που δεν συμφωνούσα και τα είπα και με την κυρία Τάισεν, ούτε και εκείνη συμφωνούσε με μένα, αλλά τι να κάνουμε, πειθαρχούμε. Είναι μια νόητη πρόταση τα βάζουμε όλα σε ένα καλάθι και τα ανακατεύουμε. Δεν είναι ωραίο. Στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας για 185 χώρες έχουν 50 υπαλλήλους. Εμείς έχουμε 87 για 27 χώρες. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή που δίνουμε προς τα Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα που δεν βλέπουμε. Αλλά και ποιο είναι επίσης το άλλο πρόβλημα. Είναι η ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Λέμε ότι πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι χώρες. Μα είναι μια ευρωπαϊκή υπηρεσία. Εντάξει, εννοείται κάθε χώρα μπορεί να έχει το δικό του στέλεχος, αλλά να το λάβουμε υπόψη μας αυτό, ότι δεν πρέπει να έχουμε τόσο πολύ γιατί είναι σαν να επιστρέφουμε στην επανεθνικοποίηση, άμα θέλει ο καθένα να είναι εκεί οπωσδήποτε παρόν και να εκπροσωπείται. Όλοι μπορούν να εκπροσωπούνται εκ περιτροπής, για παράδειγμα, κάθε δύο χρόνια. Χτες ήμουν με τον κύριο Βεζεντίνη. Οι εργαζόμενοι έχουν το Ευρωπαϊκό Συνδικάτο, την Συνομοσπονδία, μπορούν να είναι 10, από τρει-τέσσερι χώρε και να γίνεται μια εκπροσώπηση εκ Λύση μπορεί να βρεθεί. Τα λέω όλα αυτά για να τα σκεφτείτε για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαντέρ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε να ανταλλάξετε απόψεις μαζί μας σήμερα. Είναι αλήθεια ότι είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουμε οικονομικές δυσκολίες και ο καθένας αναρωτιέται δεδομένου του περιορισμού των κονδυλίων τι θα γίνει τελικά με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και τίθεται και το ερώτημα γιατί να έχουμε τόσο πολλούς οργανισμούς. Εγώ πάντως θέλω να χαιρετήσω το έργο των οργανισμών αυτών Πήγαμε στο Μπιλμπάο, εγώ έχω πάει και στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα είμαι εισηγήτρια. Συνεργάζομαι με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Καλβέ Σαμπόν κύριος. Εγώ είμαι εισηγήτρια για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Λοιπόν, πραγματικά θέλω να υπογραμμίσω το έργο σας, γιατί πιστεύω ότι γίνεται πραγματικά πολύ καλά. Το πρόβλημα είναι όμως πόσο προβάλλονται αυτοί οι οργανισμοί, πόσο γνωστοί είναι. Και δεδομένου ότι σήμερα ακόμα περισσότερο από ποτέ πρέπει να δείχνουμε στους πολίτες τι κάνουμε, πιστεύω ότι θα έπρεπε να προβληθεί περισσότερο το έργο των οργανισμών μας. Πρέπει να τους δώσουμε τα μέσα ώστε να κάνουν καλύτερη ακόμα επικοινωνία και να προβληθούν. Είναι μια αναγκαιότητα αυτό. Μια άλλη είναι να υπάρχει καλύτερη συνεργασία, με καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Αν κατάλαβα καλά αυτά που μας είπατε, η αξιολόγηση λέει ότι ακόμα κι αν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ευρύ, μεγάλο, εγώ αγωνίστηκα σε αντίθεση με τον συνάδελφο, αλλά τέλο πάντων τώρα έχουμε καταλήξει να υποστηρίζουμε το ίδιο πράγμα, να μιλάμε για μια τριμερή δομή με εκπροσώπους από όλες τις χώρες μέλη. Είναι σημαντικό, πιστεύω εγώ. Προκειμένου όμως να έχουν καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, θέλουμε παρουσία εκπροσώπων και από άλλους οργανισμούς μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, των οποίων ε, εξετάζουμε τώρα προς αναθεώρηση τον κανονισμό. Πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύουμε, γιατί έτσι θα υπάρξει καλύτερη συνεργασία και δεν θα υπάρξουν επικαλύψεις. Το είπατε και εσείς ότι χρειάζεται μια πιο καλά διαρθρωμένη συνεργασία. Τέλος, ειλικρινά, το λέω από την αρχή. Από τότε που αρχίσαμε να δουλεύουμε για την αναθεώρηση των κανονισμών των οργανισμών. Λυπάμαι για την επικάλυψη, για την κακή επιλογή ημερομηνιών, γιατί κάνουμε τη δουλειά μας, κάνουμε την αξιολόγηση και εσείς από τη, το δικό σας, τη δικιά σας την πλευρά κάνετε το δικό σας το έργο, να το έχουμε υπόψη μας ε, στο μέλλον όμως. Και αν οι οργανισμοί μεταξύ τους συνεργαστούν καλύτερα, αυτό θα ήταν κέρδος για όλους. Και εμείς πρέπει να δίνουμε πρώτοι το παράδειγμα, άρα να συντονίζουμε καλύτερα το χρονοδιάγραμμα από ό,τι το κάναμε μέχρι τώρα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Γιονγκέριους. Και μετά εσείς θα απαντήσετε. Η κυρία Γιονγκέριους πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Είναι η πρώτη φορά σε αυτή την επιτροπή, έτσι. Είναι ειδική μέρα σημερινή για την Επιτροπή μας. Γι' αυτό μπορεί να έχει αδειάσει κάπω η αίθουσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακολούθησα κι εγώ τον τριμερή διάλογο. Ακούω τα όσα λέγονται. Και εδώ ακούω μια ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση του έργου του οργανισμού σας. Των οργανισμών μάλλον αυτών. Και χαίρομαι για το αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία που απασχολούν αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, για παράδειγμα. Δηλαδή άρχισε τόσο πολύ αργά ο τριμερής διάλογος. Πώς συσχετίζεται με αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης και το έγγραφο εργασίας που θα έχουμε αργότερα. Μπορεί να πείτε πως ε, πως είμαι προληπτική. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα η συγχώνευση των οργανισμών. Η εντολή ήταν ένα χρόνο. Η περίοδος ήταν ε, ένα έτος. Πρέπει να ετοιμαστούμε για αυτή την τάση στην επόμενη θητεία. Υπάρχει δηλαδή κάποιο στον αέρα αυτό το δεχόμενο. Συμφωνώ με την αξιολόγηση των αξιολογητών ότι το κόστος της συγχώνευσης και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση αλλά και πολύ συχνά είναι υψηλότερο από το όφελος. Δεν ξέρω αν εμείς πρέπει να το αποκλείσουμε για το μέλλον, του συγχώνευση. Αυτό είναι ένα ζήτημα πάντως στη συγχώνευση. Και το άλλο είναι το εξή. Σωστά λέτε πως όταν έρθει η Επίτροπος, η Επίτροπος μάλλον ε, εδώ στην Επιτροπή μας, τότε θα έπρεπε να δούμε κατά πόσο χρηματοδότηση της εργασιακή αυτή υπηρεσία, του οργανισμού αυτού για την εργασία, να μας τα εξηγήσει, να μας πει ποιος είναι αυτός ο προπολογισμός για να δούμε τελικά τι συμφέρει. Αν συμφέρει συγχώνευση ή όχι. Για να δούμε. Είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν στον τριμερή διάλογο για το στορινούς οργανισμούς ή μήπως πρέπει εμείς να δούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς θα αντιδράσουμε στις προτάσεις για τον ΕΛΑ. Αν το χρονοδιάγραμμα δεν είναι σωστό, ίσως κάνουμε λάθη. Και σε δύο χρόνια από τώρα μπορεί να το έχουμε μετανιώσει, δεδομένου του καλού έργου των οργανισμών. Ωραία, εσείς παρακαλώ για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω πρώτα απ' όλα στον κύριο Σαμπό. Έφυγε όμως. Συμφωνώ μαζί του για το ότι μερικές φορές ε, δεν χρησιμοποιούνται παρκώς οι οργανισμοί. Ναι. Οπότε συμφωνώ με την ενθάρρυνση αυτή που θέλει να δώσει να τους χρησιμοποιούμε περισσότερο. Όντως, ο ΕΛΑ δεν έχει και πολύ σχέση με τους ήδη υπάρχοντες οργανισμούς. Πρέπει διαφορετικά να χειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε τον νέο αυτό οργανισμό. Γίνονται συζητήσεις, πολλές μάλιστα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρώτο ερώτημα που μου θέτουν όλοι είναι με έχεις ήδη τέσσερις ε, οργανισμούς, γιατί θες ένα πέμπτο» Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται επιθός, ότι χρειάζεται να επενδύσουμε όλοι για να πείσουμε ότι ο πέμπτος αυτός οργανισμός έχει εντελώ διαφορετικά καθήκοντα. Υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις και δεν το αποκλείω καθόλου να γίνεται και πολύ lobbying κατά του νέου αυτού οργανισμού από κάποιες χώρες, από κάποιους οικονομικούς παράγοντες που χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα. Μα έχουμε τόσους οργανισμούς. Γιατί να έχουμε άλλον έναν αρχή αυτή για τα εργασιακά. Ε, συμφωνώ πάντως ότι 87 είναι πολύ. Ένα διοικητικό συμβούλιο με 87, όντω. πρέπει και εδώ να επενδύσουμε για να εξηγήσουμε γιατί χρειάζεται. Πάντως, όταν μιλάω με τους διευθυντές των οργανισμών, τους έχω δει όλους, τουλάχιστον οι τρεις λένε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πραγματικά πρόβλημα, γιατί υπάρχει το διαχειριστικό συμβούλιο που τα αποφασίζει όλα και που έχει ευρύ εντολή για τους 87. Οι 87 τι είναι. Είναι επειδή υπάρχουν οργανισμοί πριν από τη δεκαετία του 80. Και κάθε φορά που είχαμε διεύρυνση προσθέταμε άλλους τρεις. Το κράτος μέλος, τα συνδικάτα του και τους εργοδότες του. Άρα για κάθε νέο μέλος είχαμε τρία παραπάνω μέλη. Ε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Με αυτό θα κάνουμε. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του παρόντος δεν έχει καμία φιλοδοξία να το αλλάξει αυτό. Τώρα η προβολή των οργανισμών συμφωνώ απόλυτα μαζί σας κυρία Σάντερς. είναι συμπέρασμα της αξιολόγησης αυτό όντω. πρέπει να κάνουμε κάτι. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση στο έγγραφό της μετά το καλοκαίρι, ώστε να φροντίσει για την καλύτερη επικοινωνία και πιο διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανισμών. Τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά, λέει ο μιλητής, να σας πω ότι ένα ερώτημα που έρχεται ξανά και ξανά και ήρθε και από τους τρεις ευρωβουλευτές γιατί έχουμε αυτή την παράλογη διαδικασία χρονολογικά. Γιατί αυτά τα τρία πράγματα τα κάνουμε παράλληλα. Είναι κάτι που προκαλεί σύγχυση, δεν είναι και πολύ λογικό. Αν όμως κοιτάξει κανείς την αναθεώρηση των κανονισμών, εισηγητής είναι ο κύριος είναι κάτι που έχει ξεμείνει. Είναι το και νομίζω ότι είναι οι μόνοι οργανισμοί που δεν έχουν ευθυγραμμιστεί ακόμα με την κοινή προσέγγιση. Και αν κοιτάξω την πρόταση, διαπιστώνω ότι χρειάζεται αυτή η ευθυγράμμιση. Δεν έχω πάει εδώ και καιρό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η πρόταση αυτή θα διευκρινίσει πολλά όσον αφορά την καθημερινή λειτουργία και την κατανομή ευθυνών μεταξύ του ε, Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθυντή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί όντως υπάρχει σύγχυση. Ποιος κάνει τι. Έχει να κάνει και με τον ορισμό προσωπικού. Η διευκρίνηση που θα έχουμε με την αναθεώρηση των κανονισμών είναι πολύ ευπρόσδεκτη και θα διευκρινιστεί και ο ρόλος της Επιτροπής. Γιατί με το ΣΕΝΤΕΦΟ, το Eurofound και τον Όσα. μερικές φορές ψάχνουμε να βρούμε ποιος κάνει τι. Και πολλές φορές ε, απευθύνομαι στις νομικές υπηρεσίες για να μου το διευκρινίσουν. Θα είναι καλό. Κύριε Γιονκέριους, ε, φυσικά δεν μπορώ να σας προκαταλάβω τι θα κάνει η επόμενη Επίτροπη. Πάντως, ακριβώς επειδή υπάρχει τέτοια σύγχυση, επί του παρόντος δεν προετοιμάζουμε τίποτα. Και η Μαριάν Τάισεν ήταν σαφής. Δεν ξέρω τι θα κάνει η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ίδιο ισχύει και για τη χρηματοδότηση. Υπάρχει ένα κονδύλι, επιπλέον χρήματα δηλαδή, δεν τα παίρνουμε από κάπου αλλού. Και αυτά τα χρήματα τα επαναδιαθέτουμε γιατί κάποιες δραστηριότητες γίνονται από τη δικιά μου γενική διεύθυνση. Δηλαδή, παίρνουμε και κάποια χρήματα από τον αστόλο, το τίποτα δεν είναι σε βάρος των οργανισμών που υπάρχουν ήδη για να χρηματοδοτηθεί ο νέος οργανισμός. Ετοιμάζεται το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και εκεί το ίδιο ζήτημα τίθεται, το ίδιο ερώτημα. Δεν βλέπω καμία ένδειξη πάντως που να δείχνει ότι θα αλλάξει η χρηματοδότηση των υπαρχόντων οργανισμών. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρος, ε, ενδιαφέροντα τα όσα ε, ακούσαμε, ειδικά εφόσον ακούσαμε, εξεκινήσαμε τον ε, τριμερή διάλογο. Όμως πιστεύω ότι τα είπατε όλα πολύ ξεκάθαρα, αφορά την ορατότητα, την αλληλοκάλυψη, το, κάστο, το κόστος και εάν παίρνουμε αυτά τα οποία πληρώνουμε και αν ξέρουμε τι είναι αυτά τα οποία ε, πληρώνουμε. Είναι ε, ξεκάθαρο λοιπόν τι θέλουμε να αποκομίσουμε ε, από αυτά. Δεν έχουν απομείνει και πολλά μέλη ύστερα από την πολύ σημαντική μας ψηφοφορία. Γι' αυτό πιο πριν είχαμε τόσο πολύ κόσμο εδώ. Όμως πιστεύω ότι μας δώσατε τις απόψεις σας, μας παρουσιάσατε τις απόψεις σας με έναν ε, πολύ ε, ξεκάθαρο τρόπο. Και εφόσον λοιπόν ε, βρισκόμαστε ακόμα στα μισά το, τη συζήτηση σχετικά με, τις, με τους οργανισμούς αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και σίγουρα θα αποθεθούμε και πάλι σε εσάς. διότι έχει έρθει η ώρα να ε, κινηθούμε για να σκεφτούμε το πώς θα αξιολογήσουμε και θα φροντίσουμε τις συγκεκριμένες, ε, τους συγκεκριμένους οργανισμούς ή αν θα πρέπει να τους αλλάξουμε εντελώ. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ε, μπορούμε να περάσουμε και στο τελευταίο σημείο τη σημερινή ημερήσια ε, διάταξη που αφορά την παρουσίαση τη ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την ελευθερία, ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, εγγυημένη ω θεμελιώδη ελευθερία, αλλά η κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί να ωφεληθεί από την καλύτερη στέχευση των πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια ειδική έκθεση από το Ευρωπαϊκό Ελληνικό ε, Συνέδριο. Ε, έχετε έρθει ε, στο παρελθόν, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, σε παλαιότερες συναντήσεις μας για να δούμε εις βάθος τα θέματα, τους φόβους, τις δυνατότητες που υπάρχουν. Καλώς ήρθατε λοιπόν. και πιστεύω ότι ο κύριος ε, Πουφάν μπορεί να ξεκινήσει. Θα σας δώσω απευθείας το λόγο για να μας, ε, παρουσιάσει, να μας παρουσιάσετε την ε, εργαλεία και να, θυμάστε ότι υπάρχει κόσμος που ε, μας βλέπει από τους υπολογιστές τους. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μέλη τη επιτροπή απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κυρίε και κύριοι. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση γιόρτασε την πέμπτη επέτειο του ιδιωτικού κανονισμού που καθιέρωσε την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Αυτή σημαίνει την ε, δυνατότητα κυκλοφορία σε όλα τα κράτη-μέλη χωρίς καμία διάκριση με βάση την ε, εθνικότητα όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης. Το 2015 περίπου 11,3 εκατομμύρια ε, Ευρωπαίοι πολίτες σε ηλικία που είναι απασχολήσιμοι ζούσαν εκτός της ε, χώρας προέλευσής τους, ε, της χώρας εθνικότητάς τους. Αυτό σημαίνει 2,7 του συνόλου του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τους κινούμενους εργαζόμενους, 1,1 εκατομμύριο άλλαξαν κάτω μέλος το 2014. Επιπλέον, 1,3 εκατομμυρία διέσχισαν τα σύνορα για να εργαστούν σε ένα διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό στο οποίο διαμένουν. Σε τι συνίσταται η εργασία μας για αυτή την έκθεση. Στη διάρκεια αυτής της έκθεσης αξιολογήσαμε τον τρόπο με τον οποίο εγγυάται η Κομισιόν την ελευθερία κυκλοφορίας και εκτιμήσαμε την αποτελεσματικότητα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη διευκόλυνση αυτής της κινητικότητας. Από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι τον Ιούλιο του 2017 αναλύσαμε τα εργαλεία ενημέρωσης ε, της Κομισιόν για να στηρίξουμε τους εργαζόμενους που έχουν εγκατασταθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος από αυτό της πρέλεσης τους, καθώς και την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα μάλλον, της ε, ε, εργατικής της βοήθειας που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει την κινητικότητα των εργαζομένων στη διάρκεια μιας της περίοδου προγραμματισμού 2014-2020. Επίσης, επισκεφθήκαμε τις εθνικές αρχές στη Γερμανία, στο Λουξεμβρού, στην Πολωνία, στη Ρουμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξετάσαμε 23 project που είχαν ολοκληρωθεί και ε, ε, εφαρμοστεί από ε, ακούς εργαζόμενους και ολοκληρώθηκαν μαζί με το ESF ε, το, ανάμεσα στο 2015 και 2016. Επιπλέον ε, του ελέγχου κάναμε και μια μελέτη για τη λειτουργία του δικτύου ΕΟΡΕΣ και δημοσι... αναλύσαμε την ποιότητα του δείγματος των θέσεων απασχόλησης που υπάρχουν ε, όσον αφορά την κινητικότητα των θέσεων. Τι διαπιστώσαμε. Κάναμε λοιπόν... Ε, η Κομισιόν έχει φτιάξει μάλλον ε, τα μέσα Your Europe, Eures και Solvit για να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στα κράτη-μέλη που έχουν ε, ε, ε κατοικούν μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που επιθυμούν να εργαστούν σε άλλο κράτος Μάλιστα, Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πλήρες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην πράξη. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν κάθε ε, καταγγελία που είναι αντίθετη με την ελευθερία και κυκλοφορία των εργαζομένων. Πέρα από αυτό το ίδιο το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ε, λίγες περιπτώσεις έχει διαπιστώσει να μην αναφέρονται συστηματικά οι υποθέσεις αυτές, οι εργαζόμενοι έχουν συχνά προσκρούσει σε εμπόδια που αν και δεν είναι παραβάσεις των δικαιωμάτων τους, ε, παρενοχλούν την κινητικότητά τους, όπως ας πούμε η μία αναγνώριση των ε, προσόντων τους, το φράγμα της γλώσσας ή η δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιδοτικών τους δικαιωμάτων. Ε, Υπάρχει δηλαδή δυναμικό που δεν ε, το εκμεταλλεύεται κανείς. Το 2014 δύο έρευνες έχουν δείξει ότι 2,9 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες έχουν εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος μέχρι το μέσα στο 2015, αλλά ότι πάνω από ένα εκατομμύριο εξ αυτών το έκαναν στην πράξη. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει παρακολούθηση των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ε, διευκόλυνση της κινητικότητας. Μέσα στο πλαίσιο ε, αυτό τα κράτη-μέλη μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για, να, για project σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την εκπόνηση προγραμμάτων και ειδικών στρατηγικών για κινητικότητα σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Το 2013 και 2014 με την, ε, τη στιγμή της έγκρισης των ε, προγραμμάτων που εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η Κομισιόν δεν γνώριζε αν τα κατημέλη θα έφτιαχναν κάποιο ε, πρόγραμμα υπέρ της κινητικότητας των εργαζομένων. Οπότε, το κύριο, η κύρια πηγή χρηματοδότησης υπέρ της κινητικότητας των εργαζομένων είναι ε, γνωστή. Είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Κοινοτομία, το ΕΑΣΥ, το οποίο το διχειρίζεται η Κομισιόν. Έχουμε εξετάσει, όπως σας είπα, 23 projects για συνοριακά ε, με το πρόγραμμα ΕΟΡΕΣ που στηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Διαφορετικό Ταμείο διαπιστώσαμε ότι ε, πολλά, πολύ λίγα project έχουν καλά αποτελέσματα, όπως ας πούμε να έχουν ε, ε, πετύχει το στόχο όσον αφορά την απασχόληση των ε, όσων ζητούσαν εργασία. Επιπλέον δεν υπάρχει ακριβής παρακολούθηση. Το Εύρες είναι το βασικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των ε, εργαζόμενων, αλλά μεγάλο κομμάτι των εθνικών προσπαθειών δεν δημοσιεύονται επιπλέον. Έχουμε κάνει ανάλυση για αυτό το πόρταλ και είδαμε ότι δεν περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές πληροφορίες για τους ετούντες εργασία, όπως ας πούμε ε, προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιωτήτων. Σύμφωνα με την Κομισιόν, 28.934 θέσεις απασχόλησης ε, καλύφθηκαν το 2016 χάρη τη συμβουλή και τη στήριξη των συμβούλων ΕΟΡΕΣ, πράγμα που είναι μόνο το 3,7% των επαφών ανάμεσα στους ετούντες εργασία και τους συμβούλους ΕΟΡΕΣ. Επί τη βάση αυτού του ελέγχου προβήκαμε σε κάποιες ε, προτάσεις, συστάσεις. Καταρχάς, πρέπει να μετρήσουμε το βαθμό της αποτελεσματικότητας των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και να αναφέρουμε εκεί όπου υπάρχουν διακρίσεις. Ενάγκη να βελτιωθεί η συλλογή των στοιχείων για το φύση της κινητικότητας των εργαζομένων και την έλλειψη ισορροπίας στην αγορά εργασίας. Βελτίωση της αντίληψης του μηχανισμού χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των... της κινητικότητας των εργαζομένων για να εξασφαλίσουμε τη συμπληρωματικότητα και να παρακολουθήσουμε καλύτερα την απόδοση αυτών, να ενισχύσουμε την παρακολούθηση και την αποδοτικότητα της πτυχής ΕΟΡΕΣ και κυρίως όσον αφορά την ε, επαγγελματική ε, αποκατάσταση και έτσι να καταστεί ένα πραγματικό εργαλείο ε, προσλήψεων στην ουσία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, υπάρχει κάποιος ε, που θα θέλει να θέσει κάποια ερωτήματα. Όχι, απλά ε, ενημερώνεστε. Άστια, είπε η πρόεδρος. Ε, νιώθω μία πίεση εδώ πέρα να απαντήσω στα όσα μόλις υπόθηκαν. Όσον αφορά τα ζητήματα διάκρισης τα οποία αναφέρατε και ε, το αν ε, αναφέρονται οι, τέτοιες, οι υποθέσεις αυτές, ε, έχουμε το δίκτυο EQUI ε, το ε, Σώμα Ανθρωπινών Δικαιωμάτων ε, και γνωρίζετε αν αντιμετωπίζονται σε κράτη-μέλη τέτοιες υποθέσεις διάκρισης κατά υπηκόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι πολύ συχνά υπάρχει η εντύπωση ότι επειδή έχουμε να κάνουμε με Ευρωπαίους πολίτες κατά κάποιο τρόπο γνωρίζουν ε, πράγματα και αντιμετωπίζονται με ε, διαφορετικό τρόπο από ότι υπήκοοι τρίτων χωρών. Ε, ενώ και αν το Συμβούλιο ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει την ικανότητα να ε, διαχειριστεί συγκεκριμένε υποθέσει διάκριση και όσον αφορά κάποια από τα ζητήματα του EURES, η Επιτροπή αυτή έχει ασχοληθεί αρκετά με αυτά τα ζητήματα και σχετικά με το πώ θα μπορούσε να βελτιώσει τα πράγματα. Θα μπορούσατε λοιπόν να πείτε κάποια πράγματα σχετικά με τη σύστασή σα πάνω σε αυτό ιδιαιτέρως ε, σχετικά με το πώς θα μπορούν να παράσχονται καλύτερα οι πληροφορίες και αν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παρέχει ένα εύρος απασχόλησης, ένα από τα σχόλια που συχνά ακούμε σχετικά με τα σώματα απασχόλησης είναι ότι προσφέρουν πολλές προφορίες για χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας που δεν πληρώνουν, πληρώνουν καλά, όμως για υψηλά καταρτισμένους δεν έχουν ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα. Θεωρείτε λοιπόν κατά τη γνώμη σας ότι κάτι τέτοιο ισχύει και στην περίπτωση του Γιουρές ε, ε, ή ε, δεν είναι τόσο γνωστά οπότε οι εργοδότες δεν τα χρησιμοποιούν τόσο πολύ όσο θα μπορούσαν. Ίσως να υπάρξουν και άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Αυτά λοιπόν είναι ε, δύο-τρία άμεσα ερωτήματα τα οποία έτσι μου ήρθαν ε, στα γρήγορα. Ε, αλλά γενικά πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα διότι θεωρώ ότι, ότι η αντίληψη κάποιων μελών μας είναι ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να, θέλουν να μετακομίσουν και να εργαστούν, όμως ε, πολλοί από αυτούς που ενδιαφέρονται ξαφνικά βρίσκουν εμπόδια. Ε, Παρ' όλα αυτά όμως ε, πρόκειται για ένα μικρό ποσοστό, σωστά. Ε, εάν κοιτάξουμε ε, ποιοι εργάζονται σε γειτονικές χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Συμφωνώ. Ξεκίνησε μεταρρύθμιση και στο ελεκτικό συνέδριο, όπου θέλουμε να σεβαστούμε αυτή την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Η διάκριση όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες που δημοσιεύονται στις χώρες μέλη, εμείς στην έκθεσή μας γράψαμε ότι μερικές φορές υπάρχουν ε, δημοσιεύσει σε κάποιες χώρες μέλη αλλά που δεν είναι σε όλα τα δίκτυα. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αρχή τώρα εργασίας η οποία θα αρχίσει να λειτουργεί το Δεκέμβριο του 2018 και ελπίζουμε ότι επί τη ευκαιρία αυτή θα μπορέσουμε μαζί να έχουμε ένα πόρταλ που θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες Πριν έρθω στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, 30 χρόνια δούλεψα στον ιδιωτικό τομέα στη Ρουμανία. Και οργανώσαμε πολλούς διαγωνισμούς. Ρωτήσατε για τη διαφάνεια. να μην υπάρχουν διακρίσεις. Για κάθε υποψήφιο θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι προθεσμίες, γιατί ανακοινώνονται σε κάποιες χώρες οι διαγωνισμοί χωρίς να αναφέρονται οι προθεσμίες. Δηλαδή μέχρι ποια μέρα συγκεκριμένα μπορεί ο υποψήφιος να υποβάλει την υποψηφιότητά του για μία θέση. Στη Ρουμανία η εξέταση αποτελείται από δύο στάδια. Υπάρχουν τα γραπτά και μετά τα προφορικά. Κατά τη γνώμη μου, για να υπάρχει εμπιστοσύνη στην οργάνωση ενός διαγωνισμού, πρέπει όλα να καταγράφονται σε βίντεο γιατί έτσι ξέρουμε τι ερωτήσεις έθεσε η Επιτροπή που θέλει να αναλύσει τα προσόντα του υποψηφίου και ποιε είναι οι απαντήσεις που έδωσε ο υποψήφιος. Οπότε, αν υπάρχει ένσταση αργότερα στη δικαιοσύνη, υπάρχουν οι αποδείξεις. Τι απάντησε, τι ρώτησε η Επιτροπή και τι απάντησε ο υποψήφιος. Τι άλλο να σας πω. Βελτίωση της γνώσης στο Γιούρες. Είναι ο βασικός στόχος, ο μεγαλύτερος. Η χρήση του Γιούρες ποικίλει από χώρα σε χώρα. Για την κάθε ανακοίνωση. Είμαι όμως ικανοποιημένος. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα όσα γράψαμε και είπαμε στις εκθέσεις μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι πολύ καλά είχε γίνει η έκθεσή μας. Αυτή είναι η απάντησή μου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικεντρωθήκαμε στο να πέσει ανεργία. Κυρίως εδώ στην Επιτροπή μας. Οι νέοι κυρίως να έχουν δουλειά. Βέβαια αυτοί που ήταν ε, νέοι, βρήκαν δουλειά, να μπορούν να παραμείνουν σε θέσεις απασχόλησης μέχρι τη σύνταξή τους. Μετά είχαμε το Γιούρες, για ένα χρόνο, από ό,τι θυμάμαι, προκειμένου να δημιουργήσει αυτή την υπηρεσία που θα βοηθούσε τον κόσμο να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη με αξιοπρεπείς μισθούς, υπό αξιοπρεπείς συνθήκες. Ψηφίσαμε πριν από λίγο για την απόσπαση των εργαζομένων. Και θέλουμε την ελεύθερη κυκλοφορία αλλά με αξιοπρεπείς συνθήκες. Οπότε οι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε μια άνετη κατάσταση και όχι σε αντιπαράθεση με, με τους δε. Αυτό ήταν το μέλημά μας τα τελευταία δέκα χρόνια θα έλεγα μάλιστα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγχρόνως από τις χώρες μέλη αλλά και από, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μας ήρθαν ε, διάφορα. Δεν πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την κινητικότητα. Εντάξει, αποκτήσαμε το Eures, το οποίο δεν λειτουργήσε όπως είχαμε επιθυμήσει, όπως περιμέναμε. Τώρα έχουμε και τους πρόσφυγες που μας έρχονται από άλλα μέρη του κόσμου και προσπαθούμε να τους εντάξουμε στις αγορές μας. και αυτοί θέλουν να μετακινηθούν με έναν τρόπο που εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε για μας. Δημιουργούμε νέα όργανα, χωρίς όμως να καταφέρνουμε να έχουμε τα αποτελέσματα το οποίο είχαμε ελπίσει να έχουμε. Και αυτό είναι εκνευριστικό. Μήπως Θα έπρεπε να ψάξουμε αλλιώς το ζήτημα. Ας πούμε εκπαίδευση. Αν ο κόσμος είναι μορφωμένος, είναι πιο εύκολο να μετακινηθεί και να βρει δουλειά. Γιατί άμα είσαι σε μια δύναμη θέση και δεν έχεις προσόντα, δεν έχεις μόρφωση, δεν φτάνει αυτή τότε αποδυναμώνεις ακόμα περισσότερο τη θέση σου. Και μένεις ε, στο χωριό σου, στην πόλη σου, στον κλάδο σου, στη δουλειά που έχεις ήδη, αν έχεις. Κρατάς ό,τι έχεις, την ασφάλειά σου και δεν κυκλοφορείς. Οπότε έτσι έχουμε μια αγορά εργασίας χωρίς τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ο κόσμος δεν κυκλοφορεί αρκετά στην αγορά εργασίας. Δεν μετακινείται. Ωραία. Το γιούρες έχουμε, θα προσπαθήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Όμως θα πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο να μας επιτρέπει να είμαστε ανθρώπινα όντα με δύναμη, που να έχουμε δουλειές. Ρωτάω λοιπόν, το βασικό με το οποίο ασχοληθήκαμε τους τελευταίους μήνες είναι το Brexit. Και αυτό θα αλλάξει τον ε, κόσμο μας. βρίσκουμε τεχνικές λύσεις Οι Βρετανοί λένε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα είναι τα πράγματα όπως ήταν πάντα. με ταυτότητες που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε σε όλη την Ευρώπη. Παρότι όσα λέγονται. Μιλάμε για την κινητικότητα, χωρίς όμως να έχουν αλλάξει πολλά. Και μάλιστα τώρα τα πράγματα αλλάζουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή λιγότερη κινητικότητα εξαιτίας του Brexit. Ναι, ξέρω σας έχω κάνει τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη με αυτά που είπα, αλλά τέλος πάντων έχετε κάτι να σχολιάσετε επ' αυτόν. Έχετε επιχειρήματα, ελπίδα να μας δώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Τι μπορώ να σας πω για τους νέους. Έχω επισκεφθεί πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δεν θα δώσω ονόματα, αλλά όταν βλέπω τους νέους στις 10 η ώρα το πρωί ή στις 2, στις 4, στα καφενεία να πίνουν Είναι θέμα εκπαίδευσης για μένα. Ένα αγόρι και δύο κορίτσια έχω εγώ. Και ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν ένα χρόνο στο Στρασβούργο με μία τάξη από ένα σχολείο της Ρουμανίας. Ήμασταν δύο ευρωβουλευτές και εγώ. Στο τέλος της συνάντησης, αυτοί τελειώναν το γυμνάσιο, έτσι, τους είπα, για μένα, εσείς που είσαστε νέοι, πρέπει να έχετε προσόντα για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να μπορείτε να μετακινηθείτε εύκολα. Και με ρώτησαν τι πρέπει να κάνω. Ε, τους είπα, πρέπει να μιλάτε τρεις γλώσσες πρώτον. Έπειτα, να ξέρετε να χειρίζεστε τους υπολογιστές, το δεύτερο. Και τρίτον, να έχετε περάσει από την ανώτερη εκπαίδευση και να έχετε κάνει και μάστερ μάλιστα. Και μετά, με όλες αυτές τις γνώσεις, μπορείτε να ε, δώσετε διαγωνισμό και να έρθετε να δουλέψετε για μας. Σίγουρα το έψο είναι ένας δύσκολος διαγωνισμός, δεν λέω, αλλά εξαρτάται από την εκπαίδευση που έχει πάρει κανείς, από τις ικανότητές του. Δεν είναι μόνο το γιούρες. Πρέπει να ξέρεις που υπάρχουν και ελεύθερες θέσεις, έτσι αλλά υπάρχει και το θέμα των διαφορετικών γενναιών. Εγώ, που γεννήθηκα το 58, βλέπω αλλιώς τα πράγματα από ότι κάποιος άλλος που είναι 26. Στον 26χρονο πρέπει να του πω αν θέλεις να δουλέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύσκολο. Δεν είναι μόνο μια εξέταση που πρέπει να περάσεις, Πρέπει να είσαι κάθε μέρα στο γραφείο σου, να παρουσιάσεις καλό έργο. Όταν ήμουν γενικό γραμματέα στο λεκτικό συνέδριο τη Ρουμανία, ήταν πολύ σημαντικό άμα ζητούσα ένα φάκελο σε 48 ώρε να έχω κάποιε πληροφορίε και δεν μου το δίνω 48 ώρε στι 72, λέω όχι ευχαριστώ πολύ, θα το κάνω μόνο μου. Έτσι είναι. Για το Brexit δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς ποιες θα είναι οι συνέπειες του Brexit. Λυπάμαι, από πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου δεν το έχουμε κάνει. Ε, δεν κάνουμε εμείς πολιτική, έτσι κι αλλιώς. Ελπίζω πάντως γιατί τα ηλεκτρονικά συστήματα, οι πλατφόρμες στη Ρουμανία έχουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα audio και βίντεο και μπορούμε να μιλήσουμε με οποιοδήποτε θέλουμε από τις άλλες περιοχές της χώρας συγχρόνως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την Ευρώπη, όπου δεν υπάρχει ίδια κινητικότητα στην Ευρώπη, όπως έχουμε στι Ηνωμένε Πολιτείε, ας πούμε. Με ηλεκτρονικά μέσα μπορούμε να κάνουμε ε, τηλεδιασκέψεις και μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα μέσα στην ίδια μέρα. Μια διευθύντρια που λέει πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό και το άλλο, τεχνικά είναι δυνατόν να γίνουν οι αλλαγές μέσα σε μια μέρα. Με δύο κουμπιά στον υπολογιστή Όμως, δεν είναι σίγουρο ότι εδώ στην Ευρώπη μπορούμε να τα κάνουμε τόσο γρήγορα. Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς έχει ερωτήσεις. στο ελεκτικό συνέδριο, στον κύριο Πούφα. Παρακαλώ εσείς. Ονομάζομαι ε, Κράτς, ε, εργάζομαι για το τμήμα πολιτικής ε, και δίνουμε πληροφορίες στην Επιτροπή ΕΜΠΛ να φέρετε κάποιες αδυναμίες για το EURES, ιδιαίτερα όσον αφορά την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, ότι τα κράτη-μέλη δεν μεταφέρουν τις ανακοινώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέσεις εργασίας και επίσης είπατε ότι μια κοινή αρχή θα μπορούσε να τα πηγαίνει καλύτερα. Ποια θα ήταν, ποιες θα ήταν οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, εργαστεί σκληρά για αυτό και υπάρχουν πολλά ακόμα δίκτυα. Ε, τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν ε, για να επιτύχουμε τους αναγκαίους στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των κρατών μελών. Μάλιστα. Η προϋπόθεση, η όρη για τη νέα αρχή της ε, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Απασχόληση μπορούμε να συνεργαστούμε με την Κομισιόν αλλά μπορούμε και να ζητήσουμε από την ε, Κομισιόν να δημοσιεύσει όλες τις ελεύθερες θέσεις. Ας πούμε, όταν υπάρχει μια ελεύθερη θέση για κάποιον ε, μηχανικό κτηρίων ή για νομικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο που πρέπει να έχει πτυχίο μάστερ ε, νομικής, να, ξέρει πότε μπορείς να, να ξέρεις πότε μπορείς να καταθέσεις την αίτησή σου, Αλλά για μας ως Ευρωπαϊκό Θεσμό Ελέγχου είναι μια νέα ευρωπαϊκή... αυτός ο νέος θεσμός δεν εξαρτάται από εμά. Δεν μπορούμε εμείς να ορίσουμε ποιοι θα είναι οι όροι. Αυτό μπορεί κανείς να το συζητήσει με την Κομισιόν για να βρεθούν κοινέ θέσεις. Okay, uh, please take the floor. Καλησπέρα. ονομάζομαι Ντεζοντών, εργάζομαι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα εντάχει να απαντήσω σε μερικά από τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν, όμως αρχικά ε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω πώς έχει η κατάσταση. Ε, ναι, μιλάμε για ένα σημαντικό θέμα, το ξέρουμε αυτό η ε, κινητικότητα των εργαζομένων αφορά το θέμα αφορά τη δυνατότητα των Ευρωπαίων ε, πολιτών ε, εργαζομένων να μένουν όπου θέλουν και να συμμετέχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή ε, οποιοδήποτε κράτους μέλους. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε μια πολιτική, έχουμε ένα νομικό πλαίσιο και στη συνέχεια έχουμε και τα εργαλεία στη, στη διάθεσή μας. Η πολιτική όπως γνωρίζετε είναι, έχει ως στόχος να, να αποτρέψει διακρίσεις με βάση την καταγωγή. Το νομικό πλαίσιο είναι ολοκληρωμένο και το γνωρίζετε αυτό. Ε, αυτό το απόγευμα το είπατε ε, εσείς κυρία Πρόεδρε. Ε, δώσατε το, προς, το πράσινο φως ε, για, την, για τον τελευταίο συμβιβασμό σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων και Έχουμε επίσης κανονισμούς και ε, οδηγίες ε, για την κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ αυτών και ε, το URES το οποίο έκανε μια επανάσταση το 2016 χάρη στο έργο του Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου πάνω στην πρόταση της Κομισιόν και επίσης έχουμε διάφορα εργαλεία, επιτροπές, επιτροπές ειδικών από τα κράτη-μέλη, κοινωνικούς εταίρους, Έχουμε την πύλη Eures, ε, καθώς επίσης και το δίκτυο, το Eures είναι και τα δύο. Ε, έχουμε ε, διάφορα προγράμματα τα οποία λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όλα αυτά λοιπόν όπως γνωρίζετε είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, όλα αυτά παρέχουν ε, κατευθυντήριες σχετικά με το τι ε, συμβαίνει, κάνουν πρότασεις και στη συνέχεια τα κράτη-μέλη βρίσκονται εκεί για να εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες κινήσεις και προτάσεις. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και διάλογο πέρσι επικεντρώθηκε στα εργαλεία και τα διάφορα προγράμματα τα οποία έχουμε και όπως ε, θα δείτε αποδεχτήκαμε όλες τις συστάσεις σας ε, και μερικές, όχι μόνο προς την Κομισιόν αλλά και αυτές προς τα κράτη-μέλη ε, θέλαμε να δείξουμε στους ε, αναγνώστες ότι πολλά ε, έχουν γίνει. Θα ήθελα να επικεντρωθώ τώρα στο EURES και την Ευρωπαϊκή Αρχή Απασχόλησης, το EURES σχετικά με τις συστάσεις. Η πρώτη σύσταση αφορά την ενημέρωση σχετικά με τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, το Eures είναι ένα από αυτά και θα ήθελα να σας πω μια ε, πληροφορία. Το, ε, το η πύλη Eures έχει ήδη μεγάλη ορατότητα κάθε μήνα έχει πάνω από 4 εκατομμύρια ε, θεάσεις ε, και 1,5 εκατομμύρια επισκέψεις. Ε, το Eures έχει πολλούς ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι προφανώς όταν το συγκρίνουμε με άλλα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο top 3 ή το 5 όσον αφορά το, την ορατότητα, ε, τώρα όσον αφορά τη σύσταση από το ελεγκτικό συνέδριο για την καλύτερη ε, χρήση των ε, διαθέσιμων πληροφοριών και την βελτίωση των δεδομένων σε αυτές τις συστάσεις θεωρούμε ότι η πρόταση που έγινε ε, για την βελτίωση. Θα επανέλθω σε αυτό. Η τέταρτη σύσταση αφορά καλύτερε συνεργίες και αυτό ισχύει ε, για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τη κάνουμε ε, και ποια είναι τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινωνικού Ταμείου ε, και σκοπός μας είναι να έχουμε μια πιο ε, καινοτόμη πρόταση πάνω σε αυτό αφού συζητηθεί το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και επίσης υπάρχουν προτάσεις για στην ε, πύλη ε, γιουρές ε, για τις πληροφορίες που αποστέλλονται από τα κράτη-μέλη στην πύλη και πολλά από αυτά θα εξαρτηθούν από τις πληροφορίες που τα κράτη-μέλη μας στέλνουν. Όπως ε, γνωρίζετε ε, υπήρχε αυτή η επανάσταση με την ε, έναρξη σε ισχύ της νέας νομοθεσίας το 2016. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και όλα τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να στείλουν όλες τις προφορίες στο, στην πύλη. Υπάρχει η δυνατότητα να κρατήσουμε μερικά από αυτά και θα το, θα το δικαιολογήσουμε να το κάνουμε αυτό και φυσικά είναι υπάρχουν δυσκολίες λόγω κάποιων τεχνικών ε, ζητημάτων ε, για τη δημιουργικότητα του συστήματος. όμω η επίβλεψη είναι έντονη και η βούληση ε, σε επίπεδο κρατών μελών και των εταίρων μας είναι πολύ μεγάλο. Το χρονολοδιάγραμμα είναι για τον Μάιο του 19 ε, θα ε, δούμε όλες αυτές τις πληροφορίες ε, και στη συνέχεια θα έχουμε τις θέσεις εργασίας στην πύλη αυτή. Η βούληση λοιπόν ήταν του Κοινοβουλίου ήταν μέσα από το EURES να κάνουμε ένα πραγματικό εργαλείο έβρεσης εργασίας και προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε και τώρα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Απασχόλησης Εργασίας ή ε, ε, θα επανέλθω ε, τον Μάιο και θα σας πω τα πάντα για την πρόταση της Κομισιόν, όμως ακόμα έχουμε αρκετά εργαλεία, έχουμε αρκετές επιτροπές όμως ε, θεωρούμε ότι θα ήταν μια καλή ιδέα και η αναφορά ε, του ελεγκτικού συνεδρίου συνεισέφερε ιδιαίτερο σε αυτό ε, και θα ήταν καλό τώρα να, κάνουμε ένα επιπλέον βήμα προς αυτήν την μονοαπευθυντική θηρίδα για να δίνουμε πληροφορίες Καθώ επίση και πληροφορίε για επιχειρήσεις ε, ε, και θα ε, επιτρέψουμε κάτι καινούριο το οποίο θα ενισχύσει τη συνεργασία διότι η, η εθνική συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για ε, να μπορέσει αυτό το νέο σώμα να συντονίζει επιθεωρήσεις κατά τόπους ε, και επίσης όσον αφορά την δυνατότητα διαιτησίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχαμε υπόψη μας με αυτή την πρόταση την οποία κάναμε τον Μάρτιο φέτος, 13 Μαρτίου συγκεκριμένα και ευελπιστούμε ότι ε, θα έχουμε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα ε, και ε, θα χρειαστεί και αυτό διότι η βούληση είναι να, η υπηρεσία αυτή να ξεκινήσει το έργο της από τον Ιανουάριο του 19. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ κύριε Πουφάν που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, και ε, ευχαριστούμε όσους μας παρακολούθησαν από τις οθόνες τους. Αυτό σημαίνει ότι τελειώνει η σημερινή συνεδρίαση εδώ. It's a great honor and pleasure for me to be here.